Και περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι οι Φιλιππίνες. Και ως ήθιστε θα δώσω το λόγο στους συντάκτες πρώτα απ' όλα. Να πάρω το λόγο. Ο κύριος Δεγόφσκε πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ε, μπορώ να επαναλάβω πια. Είναι σαν να κομίζουμε γλάφκα εσ' Αθήνας. λέμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Μιλάμε για εκτελέσεις, ε, ε, σε σχέση με τον υποθέμενο αυτό πόλεμο κατά των ναρκωτικών. Έχουμε παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, με την κράτηση της γερουσίας του Ντελήμα. Έχουμε πάρα πολλές άλλες ε, αξιόπινες πράξεις που διαπράττονται και τα μαθαίνουμε από τις ειδήσει. Ε, ζητούμε από την απελευθέρωση ε, των ε, κρατουμένων και την εξασφάλιση δίκαιης δίκης και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει ξεκινήσει έρευνα για την κατάσταση στις Φιλιππίνες. Πραγματικά ανησυχούμε και σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις που κάνει ο πρόεδρος Δουτέρτε σε βάρος των γυναικών βλέπουμε να εκφοβίζεται ο πληθυσμός ε, και ιδίω ε, να διώκονται όσοι είναι υποστηρικτές ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, ή ενό αγροτών, οικογενειακές ενώσεις των αγροτών. Μιλάμε για πάρα πολλούς νεκρούς και Ζητούμε από την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να, ασχοληθεί σοβαρά με την κατάσταση και να την αλλάξει τα ριζικά. Αυτό ζητούμε στο ψήφισμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Νίνα Τζίλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν εγκρίναμε το Μάρτιο πέρυσι ψήφισμα για τις Φιλιππίνες, είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους 7.000 άνθρωποι. Και αυτό εξαιτία ε, του λεγόμενου πολέμου κατά των ναρκωτικών του Προέδρου Ντουτέρτε. Πόσους περιμένουμε να χάσουμε ακόμα. Επικρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το θέμα αυτό ο πρόεδρος Ντουτάρτε με συλλήψεις, με παρενοχλήσεις, με βία κατά των δημοσιογράφων και όχι μόνο. Είναι πολύ κακό αυτό για τη χώρα. Ο συνάδελφος Τζακόμο Φίλγκμπετ που ήταν γενικός γραμματέας των σοσιαλιστών που κρατήθηκε και εκδιώχθηκε από τις Φιλιππίνες την Κυριακή ενώ πήγαινε να παρακολουθήσει ένα πολιτικό κογκρέσο, επειδή ήταν επικριτικό στην προηγούμενη επίσκεψή του. Δεν είναι ένα θέμα που αφορά όμω μόνο το δικό μου το κόμμα. Σημαίνει ότι οποιοδήποτε αξιωματούχος που θα βρεθεί εκεί κινδυνεύει να συλληφθεί και μάλιστα μετά την απόφαση του Πρέδρου του Τάρτε τον προηγούμενο μήνα να αποσυρθεί από το καταστατικό της Ρώμης. Είναι απαράδεκτο αυτό. Δεν είναι δυνατό να συνεχίζουμε έτσι. Υπάρχει το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ. Μπορούμε να βγάλουμε τις Φιλιππίνες από αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τσάλς Ανόκ Πρόεδρε, πριν από ένα χρόνο είχαμε το προηγούμενο ψηφισμά μας για τις Φιλιππίνες. Η κατάσταση δυστυχώς δεν έχει αλλάξει πολύ. Ο δυνατός πρόεδρος Ντουτέρτε εξακολουθεί τον πόλεμό του κατά των ναρκωτικών. Μια εκστρατεία η οποία μέχρι τώρα έχει κοστίσει τη ζωή πάνω από 12.000 ανθρώπων. Πολλοί από αυτούς νέοι. Υπάρχουν πολλές ιστορίες κατά των αυτόχθονων, κατά των ε, ανηλίκων, με παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τον ε, προηγούμενο μήνα αποφάσισε να αποσυρθεί από το καταστατικό της Ρώμης και το ποινικό δικαστήριο. Αυτό όμως δείχνει την πορεία ενός αυταρχικού επικεφαλής ο οποίος παραβιάζει τους διεθνούς κανόνες και τη διεθνή τάξη. Τα σχόλιά του δε να κάνουν και άλλες χώρες το ίδιο, ε, καθ' άλλο παρά μας βρίσκει σύμφωνος. Επίσης, θέλει να επαναφέρει τη θανατική ποινή στις Φιλιππίνες ο πρόεδρος. Κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σχετικό για την πορεία που παίρνει αυτή η χώρα. Πάντως, αυτά που λέω ότι θα συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο μέχρι να ολοκληρωθεί η θετία του το 2022 είναι και αυτό μια τεράστια απειλή. Όλα αυτά μαζί δείχνουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα στις Φιλιππίνες υπό τον Τουτέρτε οδηγεί προς μία και μόνο κατεύθυνση που κάθε άλλο παρά όμορφη είναι. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Κύριε Τάνοκ, τώρα το λόγο έχει ο κύριος Πάιτ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρο του Τέρτο και ο πόλεμο του κατά των ναρκωτικών έχει οδηγήσει στο θάνατο 12.000 ανθρώπων, πολλοί από αυτού γυναίκε και παιδιά. Πρόκειται για μαζική παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει παρενάχληση στου ακτιβιστέ, οι δράσει του Ντουτέρτε είναι σε βάρο των αυτόχθων, των μειωτήτων κλπ και από την άλλη μεριά υπάρχει και η απαράδεκτη συμπεριφορά του ίδιου του Ντουτέρτε που ζητάει τη βία, που παραβιάζει τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Νόμο. Οι απειλές του, ο εκφοβισμός, η βία πρέπει να σταματήσουν. Είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό που αποφάσισαν οι Φιλιππίνες να αποσυρθούν επίσης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και γιατί, γιατί προσπαθεί να αποφύγει να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του η πρωτοβουλία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να ερευνήσει τα εγκλήματα αυτά κατά της ανθρωπότητας στις Φιλιππίνες είναι κάτι με το οποίο συμφωνούμε γιατί χρειάζεται. Και όσοι είναι υπεύθυνοι για τα εγκλήματα αυτά μίσους πρέπει να διωχτούν και να καταλήξουν στη δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Μπάρμπαρα Λόχμπίλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βλέπουμε ότι ζητά από την ίδια την ε, αστυνομία το πρόεδρος ε, του να ε, είναι πιο επιθετική απέναντι στους ίδιους πολίτες της χώρας που διαδηλώνουν. Έχουμε 600 άτομα που θεωρούνται συμμετέχοντες στο New και τους έχουν βάλει στη φυλακή. Μιλάμε για ακτιβιστές. Η Βικτόρια Τάουλη Κόρπους, το λέμε, ε, είναι ουσιαστικά υπεύθυνη για τους αυτοχθόνους ε, που επίσης ε, αντιμετωπίζει επιθέσεις και όλοι φοβούνται ότι μπορεί να γίνουν θύματα. Εμείς χαιρετίζουμε που και το ποινικό δικαστήριο το διεθνές ξεκίνησε μια προκαταρκτική έρευνα για να δει τι γίνεται στο πλαίσιο του πόλεμου, πολέμου που έχει κηρύξει ο Ντουτέρτε κατά των ναρκωτικών, αν πρέπει να θεωρηθεί πόλεμος κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας αυτά τα οποία γίνονται στο όνομα αυτού του πολέμου. Πρέπει να διορθωθούν ε, οι πολιτικές. Ε, υπάρχουν κάποιες ανησυχητικές μελέτες για τη μελλοντική συμφωνία με τις Φιλιππίνες ε, σε ό,τι αφορά τη μη συμπερίληψη στο μέλλον της ρήτρα για τα ανθρωπιστικά δικαιώματα. Αυτό θα ήταν ένα καταστροφικό σφάλμα. Κυρία Μάλστρον, ελπίζω να το λάβετε αυτό υπόψη σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ουρμπάν Κρέσπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το, το λένε πόλεμο κατά των αγροτικών και στις ε, Φιλιππίνες δολοφόνησαν πάνω από 12.000 και με την πρόφαση του αγώνα κατά ε, της τρομοκρατίας έχουν ε, καταστήλει, έχουν δολοφονήσει όποιους είναι στην αντιπολίτευση ε, και πρόκειται για την ασιατική χώρα όπου οι περισσότεροι ακτιβιστές για το περιβάλλον έχουν σκοτωθεί ένας το 17 και οι περισσότεροι στο Μιντανάο την ε, πρωτεύουσα της εξωτερικής βιομηχανίας της χώρας και γιατί έχουν ε, καταγγείλει το στρατιωτικό νόμο της ε, διώξης όλους τους αντιπολίτες τους κατηγορούν για τρομοκρατία για την στρατιωτικοποίηση της περιοχής οπότε και κατά σύμπτωση οι ευχαριστούν την κυβέρνηση για την προστασία του. Θα πρέπει να απαιτηθεί να σταματήσει το εμπόριο όπλων, να υπάρχουν οι παραστατιωτικοί, γιατί όλοι αυτοί ε, τελικά ωφελούνται από το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και όλα αυτά θα πρέπει να παγώσουν. Να δείξουμε αλληλεγγύη, να στηρίξουμε το λαό της χώρας και συγκεκριμένα τον κόσμο που μένει στο Μιντανάο. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα τις πολιτικέ ομάδες για το ΕΛΚ και Η κατάσταση στις Φιλιππίνες προβληματίζει βαθιά γιατί έχουμε μακρύνες ε, σχέσεις αλλά και η Ιρλανδία η χώρα μου έχει σχέσεις με τις ε, Φιλιππίνες επί αιώνε έχουμε πάει εκεί έχουμε βοηθήσει τη χώρα τη εκπαίδευση. θα πρέπει να βοηθήσουμε να υπάρξει σταθερότητα και κράτος δικαίου έγινε μια ακύρωση σύμφωνου συνεργασία και είπαμε ότι είμαστε προσιλωμένοι στο κράτος δικαίου, στην οικονομική ανάπτυξη, ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Οπότε μας προβληματίζουν βαθύτερα αυτά τα οποία γίνονται. Και έχουμε όλα αυτά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος και έχουμε και γενοκτονία. Επομένως επήγει το πράγμα. Η κατάσταση είναι πολύ μεταβολή θα πρέπει να αναθεωρήσει η κυβέρνηση και θα πρέπει να αναθεωρήσει επίσης τις ληφθήσεις αποφάσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα για τους σοσιαλιστές ο κύριος Ασής έχει η κατάσταση επιδεινωθεί και η κυβέρνηση μετήλθε παν μέσων για να φημώσει την κοινωνία. Μία από στρατηγικές είναι το να ποινικοποιεί τη συμπεριφορά των ακτιβιστών, των οργάνωσεων της κοινωνίας και για αυτή την νομοθεσία έχει θεωρηθεί τρομοκράτης ακόμα και ο ειδικό εισηγητής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο κ. Σταλαβέλη. Ε, βεβαίως και όλα αυτά αποτελούν κίνδυνο ζωής και άρα θα πρέπει η πολιτική του Ντουτέρντε να αναθεωρηθεί να σταματήσουν οι δολοφονίες ηθαγενών και μελών της αντιπολίτευσης. 41 ακτιβιστές έχουν δολοφονηθεί. Θα πρέπει να λάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, και τώρα για το ΙΕΝΕΦ, κύριε Σαφχάζη. Αγαπητοί συνάδελφοι, ποιο είναι υπεύθυνο για αυτή την κατάσταση, αυτό που τη δημιουργεί ή αυτό που την αφήνει να συνεχίζεται. Το ίδιο συμβαίνει και για εμά, όπου φέρνουμε χιλιάδε εκατομμύρια πρόσφυγε σε περιοχέ που ήδη είναι περιοχέ ε, εμπορίου ε, ε, χωρίς υφές ζώνες μετά από δεκαετίες ε, ε, διαφθοράς οι Φιλιππίνες ε, που γνωρίζω πάρα πολύ καλά έχουν μετατραπεί σε μια χώρα όπου η τοξικομανία είναι δυνική. Άνθρωποι του οργανωμένου εγκλήματος είναι αυτοί που δίκουν και ο πρόεδρος προσπαθεί να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου και να σώσει τον πληθυσμό του με το 80% να τον ακολουθεί και να τον στηρίζει. Αυτές οι μέθοδοι είναι σοκαριστικές και εμένα με σοκάρουν, αλλά όχι περισσότερο από ότι οι βομβαρδισμοί στο Ιράκ, στη Λιβύη, το, στην εφεύρεση της υπόθεσης Σκρίπαλ κατά της Ρωσίας ή την δίθεν έβρεση χημικών όπλων για να βομβαρδίσουν ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Σας ευχαριστούμε κυρία Σαφχοζέλ. Η κυρία Σωράγια έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ενδιαφέρον, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να εστιαστούμε ε, στο συγκεκριμένο ψήφισμα για τις Φιλιππίνες. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Φιλιππίνες είναι εξαιρετικά ανησυχητική και μάλιστα εδώ και καιρό. Οπότε προβληματιζόμαστε ιδιαίτερως για την περίπτωση του κυρίου Φίλιμπεκ, αναπληρωτή Γενικού γραμματέα του Σοσιαλιστικού Κόμματο που συνελήφθη και δεν του επιτράπει είσοδο στη χώρα. Επίση, είναι συγκλονιστικό ότι ακτιβιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αρχηγοί αυτόχθων πληθυσμών, ακόμη και υπάλληλοι των Ηνωμένων Εθνών, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι όπω η Γερουσιαστρία Ντελήμα, βρίσκονται στο στόχαστρο τη κυβέρνηση του Τέρτε. Και φυσικά καταδικάζω δρυμύτατα τη χρήση βίας από τον πρόεδρο του Τέρτε και τα πολύ βία σχόλια που έχει κάνει βάρος των γυναικών. Και αυτός ο υποτιθέμενος πόλεμος κατά των ναρκωτικών έχει μετατραπεί σε πόλεμο κατά των γυναικών. Ε, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Είναι και καινή ώρα και είναι καθήκον μας και υποχρέωσή μας να αναλάβουμε αυστηρότερες δράσεις ε, και ακόμη αυτό σημαίνει θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τα προνόμια του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων ε, του ενισχυμένου. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Το λόγο έχει πρώτο ο κύριος Μπόγκταν Σντρογεύσκη. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω τη διαμαρτυρία μου ε, για τα σχόλια που ακούσαμε ότι μπορεί κανείς να επαναφέρει το κράτος δικαίου παραβιάζοντας το κράτος δικαίου. Αυτό όμως δεν είναι σωστός δρόμος. Αυτός είναι αδικοπραξία. Επίσης, ε, πολύ συχνά στα ψηφίσματά μας μιλούμε για απόμακρες χώρες, Βενεζουέλα, Κολομβία, Φιλιππίνες. Ερωτώ, γίνεται καμιά παρακολούθηση των ε, ε, δραστηριοτήτων μας. Γίνεται ένα follow-up, παρόλο που ε, εγώ δεν είμαι υπέρμαχος της ε, ενασχόλησης με τέτοια θέματα, αλλά μερικές φορές έχουμε πληθωρισμό στα θέματα αυτά. Θα πρέπει να προσπαθούμε και να μεριμνούμε να μην έχουμε μόνο προληπτικό χαρακτήρα τα ψηφίσματά μας, αλλά και ουσιαστικό. Να δίνεται μια συνέχεια και να δούμε αν έχουν πιάσει τόπο αυτά που λέμε. Θα πρέπει να δούμε αν όντως ε, βοηθούν τελικά κάπου αυτά τα ψηφίσματα στις χώρες στις οποίες αναφέρονται. Ευχαριστώ κύριο Ζαν Ντενανό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως, παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας, μας απασχολούν οι πολλαπλοί φόνοι που γίνονται στα πλαίσια του πολέμου κατά των ε, ναρκωτικών. Και ο κύριος ε, Ντουτέρτε ε, μένει αμετάκλητο στην εχθρική συμπεριφορά το απέναντι στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και παραβιάζει το κράτος δικαίου, έχει επαναφέρει την ε, θανατική ποινή, ε, καταπιέζει τις μειονότητες, ε, παρενοχλεί την κοινωνία των πολιτών, επιτίθεται λεκτικά απέναντι στις γυναίκες. Μάλιστα έχει ζητήσει ακόμη και το βιασμό και τη δολοφονία των γυναικών. Αυτό πραγματικά είναι απαράδεκτο, γι' αυτό και θα πρέπει να ζητήσουμε εντόνω το τέλος αυτών των παραβιάσεων και να υπενθυμίσουμε στην κυβέρνηση των Φιλιππινών τις ε, διεθνείς δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει. Ε, ο αποκλεισμό από, ε, από, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πριν το τέλος της θητείας, αλλά και άλλες ακυρώσεις οικονομικού τύπου, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να θεσπιστούν εις βάρος των Φιλιππίνων. Ευχαριστώ κύριο Συνότης Μαριάς. Το χτύπημα των εμπόρων ναρκωτικών πρέπει να γίνει στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και να επιβληθούν φυσικά αυστηρές ποινές και να μην υπάρχει καμία απόλυση από τις φυλακές των εμπόρων ναρκωτικών οι οποίοι καταδικάζονται με οποιοδήποτε πρόσχημα γιατί αυτό συμβαίνει πολλές φορές. όμως στις φιλιππίνες ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών έχει εξελιχθεί πλέον σε μια εκαθαριστική επιχείρηση που διεξάγουν οι ένοπλες δυνάμεις με πάνω από 20.000 θύματα και με εξοδικαστικές εκτελέσεις. ταυτόχρονα ο πρόεδρος των φιλιππίνων αξιοποιεί αυτή την ευκαιρία του πολέμου όπως λέει κατά των ναρκωτικών για να αντιμετωπίσει πολύ σκληρά τους πολιτικούς του αντιπάλους και φυσικά οδηγεί τις φιλιππίνες σε ακραίες καταστάσεις με βία κατά των γυναικών και επαναφορά της θανατικής ποινής. επομένως πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά των φιλιππίνων όπως είναι να καταργηθούν οι γενικές δασμολογικές προτιμήσεις της ευρωπαϊκής ένωσης με τις οποίες εισάγονται πλέον αδασμολόγητα προϊόντα των Φιλιππίνων εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Ιγνάσιο Κοράο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το κλίμα τρόμου που επικρατεί στις Φιλιππίνες είναι πολύ ανησυχητικό. Δεν μπορούμε πια να το ανεχόμαστε. Ο σκληρός πόλεμος ενάντια στα ναρκωτικά του Πρόεδρου του Τάρτε έχει οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό θυμάτων που πέφτουν ε, με τα χτυπήματα, από τα χτυπήματα της αστυνομίας ή των πληρωμένων στρατιωτικών. Ε, Θα ρίνεται η ένοπλη καταστολή των ακτιβιστών και των γυναικών. Αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Ε, βέβαια, η καταπολέμηση των εμπόρων ναρκωτικών είναι ένας στόχος ε, τον οποίο μπορούμε να συμμεριστούμε. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με εξοδικαστικές διαδικασίες από πλευράς της ε, μισθοφορικής αστυνομίας. Ε, ε, επίσης φαίνεται ότι χτυπιούνται τα πιο, φτωχά, πιο φτωχές περιοχές και γειτονιές της Μανίλα. Πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε κάθε δυνατή πίεση στο, απέναντι στον πρόεδρο του Τάρτε, ώστε να υπάρξουν δίκαιες δίκες για αυτόν τον μακρύ κατάλογο υπόπτων. Σας ευχαριστώ κύριε Στάμπα Σόγκορ. Ευχαριστώ. Ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών στις Φιλιππίνες έχει επεκταθεί και σε άλλα θέματα που μας επισημαίνουν οι οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, ε, το κρατικό μονοπόλιο της καταστολής ε, είναι ανησυχητικό, γιατί μόνο το κράτος, οι αρχές επιβολής του νόμου χρησιμοποιούν αυτό το μηχανισμό της καταστολής αλλά έχουμε και κάποιους βιζιλάντες, κάποιες ομάδες φρουρών που ε, αυτοδικούν, να αναλαμβάνουν την δικαιοσύνη στα χέρια τους με την ανοχή του κράτους. Έτσι καταπατώνται τα δικαιώματα των πολιτών για ασφάλεια και προστασία που κανονικά θα πρέπει να εξασφαλίζονται από την αστυνομία. Μας ανησυχεί αυτή η έλλειψη ασφάλειας στις Φιλιππίνες δεν είναι δυνατόν να επιτρέπονται εξοδικαστικές εκτελέσεις. Είναι σαν να γυρίζουμε σε βαρβαρότητες προϊστορικές, λόγω της έλλειψης κανόνων. Μόνο ένα δικαστήριο θα πρέπει να αποφασίζει αν κάποιο είναι ένοχο και να επιβάλλει κάποιε ποινέ. Όλα αυτά είναι απόρρια τη κυβερνητική πολιτική του κ. Ντουτέρτε. Σα ευχαριστώ. Κύριο Φάμπιο Καστάλντο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν εμποδίζουν τη δικαιοσύνη, ε, πυροβολήστε τους. Αυτό έλεγε τον περασμένο χρόνο ο Ντουάρτε όταν έδινε οδηγίε στην αστυνομία πώς να επιτεθεί κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι λόγια τα οποία δυστυχώς ισχύουν ακόμα. Πάνω από 10.000 νεκροί, πάνω από το μισό από την αστυνομία έχει σκοτωθεί. Επειδή δίθεν αντιστάθηκαν στη σύλληψη. Ο υποτιθέμενος πόλεμος ενάντια στα ναρκωτικά ε, οδηγεί στην άρνηση της δικαιοσύνη χιλιάδες αθών και οικογενειών τους. Ε, η καταπολέμηση αυτής ε, της ε, σε Λίγοι ακτιβιστές, δημοσιογράφοι και πολιτικοί ε, αντιστέκονται ακόμα, ενώ όσοι συλλαμβάνονται ε, ε, καταδικάζονται χωρίς δίκη και χωρίς αιτιολογία. Ακόμα και μια γερουσία από η οποία συνελήφθη υπέστη την ίδια διαδικασία άνευ δίκης. Διεθνές δικαστήριο. Έχουμε φτάσει στο Διεθνές δικαστήριο για να πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε μόσο ώστε να υποχρεώσουμε τις Φιλιππίνες σεβαστούν τι διεθνεί του δεσμεύσει και να σταματήσει ο πρόεδρο έρτε να δράμα αυτή την πολιτική τρόμου. Σα ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τη διαδικασία Κατσδιά και στρέφουμε και πάλι στην Επίτροπο, την κυρία Σεσίλια Μάουστρομ για την τελική τη ομιλία για το θέμα αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε εκφράσει τι έντονε ανησυχίε μα για τα ζητήματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στι Φιλιππίνες αρκετέ φορέ και σε διμερεί ε, συναντήσει σε διάφορα πολιτικά επίπεδα αλλά και με τη μορφή δηλώσεων. Αυτά τα ζητήματα που ετέθησαν εδώ, ο ψηλό αριθμό ε, των ε, δολοφονιών ε, εξ ονόματο εκστρατεία κατά των ναρκωτικών, η ατιμορρησία, η απόσυρση από το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο, η επανεισαγωγή τη θανατική ποινή αλλά και η μείωση του όριου ηλικία στην ποινική ευθύνη στα 19 χρόνια. Πέραν αυτού, Έχω τεθεί θέμα υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη σύλληψη του γερουσιαστή Λίμα και ε, περιορισμό τη ελευθερία τη έκφραση, αλλά και θέματα ε, περί ε, μία ανεξαρτησία των θεσμών και της δικαιοσύνη. Αυτά τα θέματα έχουν τεθεί ήδη σε διάφορες δηλώσεις στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με δηλώσεις της ΥΠΑ της εκπροσώπου και αναφέρονται εκτενώς στην έκθεση παρακολούθησης των ε, G20 συν. Ε, εγώ προσωπικά σε πολλές περιπτώσεις συναντήθηκα με αξιωματούχους της κυβέρνησης των Φιλιππίνων και εξέφρασα αυτές τις ανησυχίες μας. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ε, καταγγελία της 21ης Φεβρουαρίου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου κατηγορούνται 260 άτομα ότι ανήκουν στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Ε, ο ειδικό εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών έχει ε, αναφερθεί στο θέμα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των αυτοχθόνων. Και επίσης σε ό,τι αφορά όλα τα άτομα που βρίσκονται σε αυτόν τον κατάλογο, αναμένεται η κυβέρνηση των Φιλιππίνων να ακολουθήσει τις νόμιμες ε, διαδικασίες ε, που απορρέουν από το εθνικό και διεθνές δίκαιο και να σέβεται το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και να διασφαλίζει την προσωπική σωματική τους ακαιρεότητα και ασφάλεια και να εγγυηθεί μια δίκαιη δίκη για όλα αυτά τα άτομα. Οι απελάσεις επίσης έχουν ε, τεθεί από τον ε, ως θέμα από τον Τζάκομο Φιλιππέτη. Καθώς επίσης και οι διάφορες παρόμες πολιτικές δραστηριότητες. Όπως ξέρετε, κλήθηκε να συμμετέχει στη συνεδρίαση ενός κόμματος το οποίο ε, είναι τόσο μέλος της Γερουσίας όσο και του Κοινοβουλίου και κρίθηκε παράνομο απελάθηκε από τη χώρα για πολιτικούς λόγους ε, κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής εδώ της κυβέρνησης. Έχουν γίνει εξοδικαστικές ε, εκτελέσεις και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό στις ε, Φιλιππίνες σύμφωνα με την έκθεση Sin. Τόσο οι Φιλιππίνες όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πολλά να κερδίσουν από την ε, δημιουργική συνεργασία. Η Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία ε, τέθησε ισχύ την 1η Μαρτίου αυτού του έτους και προβλέπει έναν διαρθρωμένο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ των συμβαλόμενων μερών που θα ασχοληθεί με όλα τα ζητήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναφέρθηκαν οι διεθνείς δεσμεύσεις από πολλούς από εσάς που αναφέρονται στην έκθεση Sin. Τον Ιανουάριο ήδη τονίσαμε ότι υπάρχουν αρκετοί τομείς στους οποίους έχει σημειωθεί πρόοδος από την κυβέρνηση των Φιλιππίνων. Για παράδειγμα ισότητα των φύλων, υγεία, εκπαίδευση, εργατικά, κοινωνικά δικαιώματα, καταπολέμηση της διαφθοράς και προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο ε, φάνηκε στην ε, έκθεση ότι οι εξοδικαστικές εκτελέσεις ιδιαίτερα εξ ονόματος του πολέμου κατά των ναρκωτικών έχουν οδηγήσει σε ατιμορρησία. Επίσης αναφέρθηκε και η επανεισαγωγή της θανατικής ποινής. Προσωπικά ήδη έχω εκφράσει τις ανησυχίες μας ε, στον ε, αρμόδιο υπουργό και του ε, έχω επισημάνει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Παρακολουθούμε λοιπόν στενά τις εξελίξεις και φέτος η αποστολή παρακολούθησης JSPC θα εστιάσει σε ζητήματα που αφορούν τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προβεί σε αξιολόγηση των εξελίξεων προτού σκεφτεί ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΕ θα συνεχίσουν να πιέζουν για αυτά τα ζητήματα με τρόπο επικοδομητικό και σαφή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Έξι σχέδια ψηφίσματο έχουμε λάβει κατά τα ολοκλήρωση της συζήτησης από το ΕΛΚ, από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, το σχέδιο ψηφίσματος το ECR, το σχέδιο ψηφίσματο από τους Φιλελεύθερους από τους Πράσινους, καθώς και ένα σχέδιο ψηφίσματος από την ΓΚΟΕ. Ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτηση για το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία θα γίνει